Uh, dear colleagues, good morning. I hope that we can begin. Ο πρόεδρος, ελπίζω ότι είμαστε στη θέση να ξεκινήσουμε. Και ελπίζω να είναι συναρπαστική η ψηφοφορία και να μην έχουμε θέματα. Ναι, ναι, ζήτησα, ζήτησα, να έχουν περισσότερη ζέστη. Εδώ και μισή ώρα το ζήτησα. Αλλά δεν βλέπω τα αποτελέσματα από τη θερμοκρασία του δωματίου της αίθουσας. Okay, So, I hope you have your voting cards ready. Ελπίζω έχετε τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.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 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθυμών 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 2 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος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 εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 1 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 2. Έντεκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο της εκθέσεως. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια κυρία Ράντιεφ. Και τώρα η έκθεση του υποφαινομένου όσον αφορά την παραγραφή για τα τροχέα. Υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ τη τροπολογίας 10. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον υποφαινόμενο. Πάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Μαστάλκα προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ Α, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. τρία Υπαριθμών τρία, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. έξι Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για 14 μιλάω. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του σχεδίου γνωμοδότησης το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μαστάλκα. Πάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Λεμπρετών εφαρμογή των διατάξεων συνθήκες όσον αφορά, συνθήκες όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Μία ε, ψηφοφορία κάνουμε ηλεκτρονικός, έναρξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, Μία ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Γκούτελαν για τις διασυνοριακές ανταλλαγές. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Είναι το σημείο 26 της ημερήσιας διάταξης. Διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ Ένωσης και Τρίτων χωρών Shall I read out the whole title? Item 26. Item... Να διαβάσω το, όλο τον τίτλο. Το 26. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Άντερσον. Για το σημείο 27 της ημερήσιας διάταξης, έναξη ψηφοφορίας για την έκθεση του κυρίου Άντερσον. Uh, adopted Εγκρίνεται. Κύριε Άντρισον, συγχαρητήρια. And we have a second, Mr. Έχουμε μία ακόμη έκθεση του κυρίου Άντερσον. Επιτρεπόμενες χρήσεις έργων κλπ. κλπ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια κύριε Άντερσον. Μία ακόμη έκθεση της κυρίας Γούτελαντ. Α, έχει αναβληθεί η ψηφοφορία αυτή. Με ενημερώνουν. Ναι. No, somebody else did not cover that. must be postponed. Yes. Mr. Cavada asked for that to be postponed yesterday. Do we want Mr. Mr. Foss. Κύριε Φως, έχετε το λόγο. Πριν φτάσουμε στο σύστημα εισόδου-εξόδου, αυτό είναι το επόμενο σημείο, γιατί γι' αυτό θέλω να πω κάτι. we, postponed yesterday. Μα το αναβάλαμε χθε από τη συζήτηση του σημείου 10. that this is this is a mistake. Πρόκειται περί σφάλματος όμως. Πρέπει να ψηφίσουμε για τη θεσπιση συστήματο συστήματος εισόδου-εξόδου. Κύριε Φώση, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, υπήρχε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και εγώ δεν ε, συμφωνώ με αυτή την πρόταση. Τουλάχιστον όσον αφορά το σημείο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας. we have the legal... Είναι εδώ η νομική υπηρεσία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Είναι σαφές, ε, κατά την άποψη της νομικής υπηρεσίας, ότι το άρθρο 77.2β ε, και το άρθρο 87 παράγραφος 2 σημείο α σε συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σωστή νομική βάση για την προτινόμενη προτινόμενο κανονισμό εισόδου-εξόδου, λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι το άρθρο 88 παράγραφος 2α δεν μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη νομική βάση, είναι ε, η εξή. Η λόγη είναι η εξή. Πρώτον, ο στόχο και το περιεχόμενο τη πρόταση ε, και βάσει τη νομολογία του δικαστηρίου. Οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με την Ευρωπόλ ε, είναι μόνο δευτερεύουσες και συγκυριακές στο πλαίσιο του προτινόμενου κανονισμού. Δεύτερον, λαμβανομένου υπόψη του κειμένου του συστήματος για τον κανονισμό εισόδου-εξόδου, μια σαφής διάκριση πρέπει να γίνει. Η χρήση του άρθρου 87 είναι η νομική βάση και δικαιολογείται αυτό λόγω της ανάγκης ρύθμισης της πρόσβασης του συστήματο εισοδου εισόδου-εξόδου από τι εθνικές διοκτικέ αρχέ. Αντιθέτω, η Ευρωπόλ μπορεί Ούτω ή άλλω έχει ήδη πρόσβαση στο σύστημα αυτό μέσω των διατάξεων που αναφέρονται στην σύμβαση τη Ευρωπόλ. Αυτέ οι διατάξει δεν επηρεάζονται από τον προτινόμενο κανονισμό. Ουσιαστικά, ο κανονισμό για το σύστημα εισόδου-εξόδου ορίζει απλώς τους ε, όρους πρόσβαση της Ευρωπόλ. Τρίτον, ε, το άρθρο 17 της Σύμβασης της Ευρωπόλ ήδη ορίζει ήδη προβλέπει πώς γίνεται η πρόσβαση της Ευρωπόλ στο σύστημα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η πρόσβαση και η χρήση των πληροφοριών από την Ευρωπόλ πρέπει να διέπεται από το απαραίτητο, από το κατάλληλο νομικό μέσο όπως, και θα, όπως θα ισχύσει και για τον κανονισμό εισόδου-εξόδου. Ο προτινόμενος κανονισμός δεν δημιουργεί νέα καθήκοντα για την Ευρωπόλου, ούτε αυξάνει τις ε, εξουσίες της ε, σε σχέση με το τι ε, αναφέρεται ήδη στον κανονισμό της Ευρωπόλου, ούτε τροποποιεί τα καθήκοντα όσον αφορά την αποθήκευση, τη χρήση, την ανάλυση, την επεξεργασία δεδομένων. Επίσης, η διατύπωση του άρθρου 87 και του άρθρου 88 είναι διαφορετική. Ε, μέτρα στο 87 και κανονισμός ε, ρύθμιση στο άρθρο 88. Τα μέτρα του άρθρου 88 δεν ε, συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό του, του, του συστήματος εισόδου εξόδου βάση του άρθρου 88 οι διατάξεις ε, αυτές πρέπει να ε, θέτουν και τις διατάξεις που αφορούν την εποπτεία, την παρακολούθηση ε, των δραστηριοτήτων της ευρωπόλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο δεν ισχύει στον κανονισμό του συστήματος εισόδου-εξόδου, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση, αν θέλετε, να προσθέσετε αυτή τη νομική βάση. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, να προσθέσω και το εξή, ότι σύμφωνα με νομολογία του δικαστηρίου, το να ε, προσφύγουμε, να καταφύγουμε σε διάφορες νομικές βάσεις ε, ε, μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως εξηγείται στο σημείωμά μας. Βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φως. Κοιτάξτε, αν κατάλαβα κάτι, το 88 2α δεν είναι τελικά απαραίτητη κοινωνική βάση πλέον. Ερωτώ λοιπόν, το άρθρο 88 θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε τελείως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε στην ψηφοφορία αυτή την πρόταση. Μπορούμε να το αναβάλουμε αν δεν μπορεί να πάρει θέση αυτή τη στιγμή η νομική υπηρεσία. Μήπως πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ναι, υπάρχει σύγχυση. Εγώ έλεγξα στα έγγραφά μου. Όντως, ο κύριος Καβαντά ζήτησε αναβολή. Και από την αρχή είπαμε ότι το σημείο αυτό αναβάλλεται. Βλέπω λοιπόν ότι επειδή δεν είναι σαφής η θέση μας, προτείνω όλη η ψηφοφορία να αναβληθεί. Uh, uh, Συνεχίζουμε λοιπόν με την έκθεση Γιούταλα, αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Ο κύριος Ζάγερ. Ευχαριστώ. Ναι. Δεν έχουμε όμως το κείμενο και τον κατάλογο ψηφοφορίας για την έκθεση αυτή. Προτείνω λοιπόν να αναβληθεί και αυτή η ψηφοφορία. Λοιπόν, επί ποιου κειμένου ψηφίζουμε. Πρόκειται για την εισήγηση, τη γνωμοδότηση της κυρίας Κάουταλα με ημερομηνία όπως τροποποιήθηκε εξάλλου εχθές το βράδυ Τροπολογία 6. Συμπεράσματα. Εκτός ε, λοιπόν από αυτήν την αλλαγή, δηλαδή τη λέξη could, που αντικαθιστά τη λέξη should, το κείμενο είναι ως έχει. Δεν έχετε πάρει αυτή την τροπολογία. read out, read out the sorry. I'm, uh, Ναι, είδα πραγματικά ότι δεν έχει διανεμηθεί στα μέλη της Επιτροπής ε, το κείμενο. Συμφωνείτε λοιπόν να αναβάλουμε το σημείο αυτό. Δεν έχω άλλη δυνατότητα δυστυχώς. Προφανώς η γραμματεία δεν έστειλε το κείμενο. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει ψηφοφορία. Αναβάλλεται λοιπόν η ψηφοφορία. Συνεχίζουμε με την έκθεση Τε για τον κώδικα Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Πρόκειται για μία ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κύριε Σβεύκα sorry for this misunderstanding. Και ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση που επικράτησε. Yeah, this is all for the votes. Ολοκληρώσαμε με την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Με το επόμενο σημείο πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Σβιεύκα. Το σημείο 31 της ημερησίας διάταξης που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε διαφορές γάμου και διαφορές γονικής μέρημνας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση αυτή, την οποία θα σας παρουσιάσω τώρα, είναι μία έκθεση και 24 τροπολογίες. Ελπίζω ότι θα στηρίξετε την έκθεση αυτή καθώς ε, η έκθεση αλλά και οι τροπολογίες που σας υποβάλλω ότι κατοπτρίζουν την προσέγγιση όσον αφορά την τροπολογία της, του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Ζητώ συγγνώμη. Όποιος θέλει να συζητήσει, παρακαλώ πολύ να βγει έξω. Οι υπόλοιποι καθίστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ με την γενική ιδέα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και <clears throat> όσον αφορά τις ε, τροπολογίες ε, που υποβάλλω, νομίζω ότι μπορούμε να τις ταξινομήσουμε σε διάφορες κατηγορίες και θα μπω στις λεπτομέρειες για να σας παρουσιάσω τις τροπολογίες αυτές που καλύπτουν καταρχήν κάποια κενά. Παραδείγματο χάρη στον τίτλο προσθέσαμε την περίπτωση των διεθνών απαγωγών παιδιών. Εδώ αυτό το έχουμε προσθέσει στον τίτλο. Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να προσθεθεί στο σημείο 1 του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Δεύτερη κατηγορία τροπολογιών αφορά συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κυρίως. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων όταν παραδείγματος χάρη να υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ανταλλάξουν οι αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα για ένα παιδί το οποίο είναι θύμα απαγωγής. Τώρα, για τα παιδιά αυτά που πρέπει να ανατεθούν σε οικογένειες εκτός της οικογένειάς τους, τα κράτη-μέλη του εν λόγω κράτους θα πρέπει να εξετάσουν τις περιπτώσεις ένα παιδί να τοποθετηθεί σε μια οικογένεια εκτός της δικής του οικογένειας Οι αρμόδιες αρχές ε, θα πρέπει όμως να εξετάσουν και τη δυνατότητα κάποια μέλη της ε, οικογένειας να αναλάβουν ε, το παιδί για να μπορέσει να έχει επαφή με την πραγματική του οικογένεια. Το θέμα της εκτέλεσης μιας απόφασης και της αρμοδιότητας των δικαστηρίων στο σημείο 36 νομίζω ότι βλέπετε ότι οι τροπολογίες αυτές συμπληρώνουν το κείμενο. Δεν αρκεί εδώ να υπάρχουν δηλώσεις εάν δεν εκτελείται μία απόφαση στο χρονικό διάστημα που ακολουθεί, τις έξι εβδομάδες δηλαδή που προβλέπει ο νόμος. Εάν δηλαδή δεν τηρούνται αυτές οι προθεσμίες για την εκτέλεση των αποφάσεων, προβλέπεται το δικαστήριο να ενημερώσει για την μη εκτέλεση της απόφασης και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη μη εκτέλεση. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι θα πρέπει οι προθεσμίες να είναι σαφείς, να τηρούνται όσον αφορά την εκτέλεση πάντα των αποφάσεων, γιατί αυτό είναι πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να ενδιαφέρουν τις αρμόδιες αρχές και να δίνονται από το δικαστήριο. Τώρα, τα αρμόδια δικαστήρια για τις απαγωγές παιδιών. Συμφωνώ απολύτως με τις διαδικασίες που ουσιαστικά έχουν σαν σκοπό να απλοποιήσουν τις ε, διαδικασίες που σήμερα είναι περίπλοκες, που είναι δύσκολες και θα πρέπει να βρούμε λύση που να επιτρέπει στον δικαστή, στους δικαστές οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την ουσία μιας υπόθεσης, έτσι ώστε η διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων να είναι χρήσιμες και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε να μην υπάρχει απολύτως κανένα εμπόδιο ε, όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ε, μερών. Παραδείγματος χάρη, όταν ε, αναφέρουμε αυτό το θέμα των διεθνών απαγωγών. Και θυμάστε στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε αυτού του κανονισμού, που αφορά αυτόν τον κανονισμό, που είναι δηλαδή ήδη μια αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Πάντα ε, θεωρούμε ότι το συμφέρον του παιδιού πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά ε, μιας τέτοιας διαδικασίας. Πρέπει επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τα παιδιά. Στα πλαίσια των ε, συνθήκων και βάσει της αρχής της ε, επικουρικότητας πρέπει να προτείνονται κοινέ διαδικασίες όσον αφορά την ακρόαση ενός παιδιού. Παρόλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε τα εν λόγω παιδιά να μπορούν πραγματικά να μιλήσουν έτσι ώστε η απόφαση που λαμβάνεται από το δικαστή να είναι πάντα η καλύτερη όσον αφορά την προστασία ε, των δικαιωμάτων του παιδιού. Και γι' αυτό και η οποιαδήποτε απόφαση δικαστηρίου Ιδιαίτερα αν ένα δικαστήριο αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται να ακούσει ένα παιδί, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πάντα στα πλαίσια της απόφασης να αναφέρεται γραπτός ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να ακούσει το συγκεκριμένο παιδί. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε σε μια διαδικασία, αλλά θέλουμε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται υπόψη καταρχήν το συμφέρον του παιδιού. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που θέλω να κάνω σε σχέση με τις τροπολογίες μου, σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να εξετάσουμε και τις τροπολογίες που θα υποβάλουν άλλοι ε, μέλη της Επιτροπής. Η προθεσμία για την υποβολή των ε, τροπολογιών 25 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σιεύκα, γιατί όπως πάντα μας παρουσιάσατε ένα πάρα πολύ καλά δομημένο σχέδιο εισήγησης εγώ συμφωνώ στα περισσότερα από αυτά που προτείνετε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζετε το συμφέρον του παιδιού στην καρδιά των ε, εργασιών σας. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σωστή ε, αφετηρία, αν θέλετε, για μας. Βεβαίως υπάρχουν τελείως διαφορετικές ε, καταστάσεις. Η καλύτεροι, όμως ε, επιλογή και απόφαση για το παιδί είναι αυτή που πάντα θα πρέπει να μας καθοδηγεί. Και χαίρομαι που έτσι ακριβώς λειτουργείτε. Το θέμα τώρα είναι το νωρίτερο δυνατόν το παιδί να επιστρέψει στην οικογένειά του. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει, όπως πολύ σωστά το προτείνεται, να το πετύχουμε με κάθε τρόπο. Επίσης, θεωρείται πολύ σημαντικό να ακουστεί ένα παιδί. Και αυτό θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να θέσουμε κάποια ελάχιστα ε, όρια και προϋποθέσεις και βεβαίως να διαπιστώσουμε ότι η βάση της ηλικία του κάθε παιδιού ε, γίνονται και οι αντίστοιχες διαδικασίες ακρόασης. Γιατί βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η ίδια διαδικασία, να χώρα η ίδια διαδικασία ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν με τους ε, γονείς ή έναν από τους δύο γονείς. Πάντα υπάρχουν ε, τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει καταρχήν να εξεταστεί η περίπτωση συγγενικών προσώπων ή μελών της οικογένειας που μπορούν να αναλάβουν το παιδί. Εγώ σαν αρμόδια για τα θέματα αυτά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές φορές αρμόδια άτομα που μπορούν να λάβουν υπόψη τους το πραγματικό συμφέρον του παιδιού και αναρωτιέμαι αν ε, η απόφαση που λαμβάνεται πολλές φορές ε, να απομακρυνθεί ένα παιδί από την πραγματική του οικογένεια και να το αναλάβει μία άλλη οικογένεια, θα πρέπει να δικαιολογείται πάντα από πάρα πάρα πολύ σοβαρούς λόγους. Είναι καταστάσεις ε, που πραγματικά πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή, ε, έχω πολλά ερωτηματικά και πολλές επιφυλάξεις. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για μια τέτοια απόφαση, γιατί όπως ξέρετε οι επιπτώσεις είναι πάρα, ή μπορεί να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρές. Όσον αφορά τώρα την επιλογή των δικαστηρίων, ναι, και εγώ σαν ε, ε, αρμόδια για τα θέματα αυτά, γνωρίζω την ε, παράδοση που μπορεί να προκύψει από την συχνότητα με την οποία προκύπτουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις σε ένα δικαστήριο. Η συγκέντρωση λοιπόν των υποθέσεων αυτών σε αρμόδια δικαστήρια είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Το θέμα του πόσο έγκαιρα ξεκινάει η διαδικασία διαμεσολάβησης θα υποβάλω μια τροπολογία για το θέμα αυτό και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερη βάση για να λάβει υπόψη του κανείς τα πρώτα στάδια αυτής της διαδικασίας και το πόσο νωρίς μπορεί να ξεκινήσει η διαμεσολάβηση. Βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλα τα πολύ σύγχρονα ε, είδη, αν θέλετε, οικογενειών, σύγχρονη ζωής. Το αναφέρετε αυτό, αλλά μετά στις τροπολογίες σας δεν βλέπω τίποτα από αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε βεβαίως τι ισχύει στις ε, χώρες και θα λάβω υπόψη μου αυτό, θα υποβάλω και μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεών σας. Πιστεύω ότι η πολιτική γραμμή που θα ακολουθήσουμε είναι κοινή και νομίζω ότι στις περισσότερες εκθέσεις που επεξεργαστήκαμε από κοινού είχαμε κοινέ ε, κατευθυντήριες γραμμές και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και σε αυτή την έκθεση την εξαιρετική μας συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος και είναι το λόγο στον κύριο Λεμπρετών. Να προσθέσω δύο λόγια για την έκθεση αυτή πολύ σημαντική γιατί όπως και ο κύριος Βιέφκα μας ε, τόνισε αφορά αυτού του είδους της διεθνής αγωγές των παιδιών και έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που μας ε, έχουν επισημανθεί από τους εμπλεκομένους. Θα πρέπει επομένως κάπως να βελτιώσουμε το σύστημα και ευχαριστούμε κύριε Σβιεύκα για τη δουλειά σας. Ε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τροπολογία, ακόμα δεν τη συζητήσαμε. Είναι τροπολογία υπαριθμών 6, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ε, η καταγραφή της ακρόασης του παιδιού. Και το τέλο πάντων. Οπότε και έτσι, χωρίς πίεση να μπορεί να γίνει η ακρόαση του ανηλίκου σε αποδεκτές συνθήκες, άρα είναι εύστοχη αυτή η πρόταση. Ε, επίσης, να προστατευτεί η εθνική κυριαρχία. Επομένως, ε, συμφωνεί και ο Σβιεύκα νομίζω, γιατί στην τροπολογία 2 λέει ότι θα πρέπει ό,τι αναγνωρίζεται σε κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, γίνει σεβαστό από την ρύθμιση που θα κάνουμε. Άρα θα πρέπει το εθνικό δίκαιο να συνεχίσει να ισχύει και τώρα το πιο βασικό για το θέμα μας είναι η συνεργασία αλλά να μην έχουν κάποιο είδου ε, εξομοίωση και ισοπαίδωση. Επομένω, όταν υπάρχουν κάποιε εθνικέ ιδιοτυπίε να διατηρηθούν. Σα ευχαριστούμε, λέει ο δεν βλέπω άλλος να ζητεί το λόγο. Οπότε, ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο και θα κάνουμε μέχρι τις 11 ένα διάλειμμα, οπότε και τότε θα έχουμε την ακρόαση για τις νομικές συνέπειες του Brexit.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ορίσατε στην ακρόασή μας. Το θέμα του είναι οι νομικέ συνέπειες του Brexit. Σας καλωσορίζω που ήρθατε και να ευχαριστήσουμε την κυρία Ντενούτα Χιούμπνερ, την πρόεδρο της Επιτροπής Συνεγματικών Υποθέσεων. Της δίνουμε το λόγο ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Επίσης, μια που έχουμε εμπλακεί ως Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία για να μπορούμε να προετοιμαστούμε και θέλουμε να ληφθεί κοινή απόφαση από όλες τις κοινοβουλικές επιτροπές. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε συνυπεύθυνοι ούτω ώστε να ολοκληρωθεί αυτή χωρίς προηγούμενο διαδρομή. Είμαστε ακόμα στην αρχή της. Και όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επομένω, εκτός από αυτή τη διαδικασία, θέλουμε να γίνουν τα πράγματα όπως είναι καλύτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους Ευρωπαίους. Γιατί αν δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την αποχώρηση, ε, θα έχουμε εντυπωσιακέ και δραματικές συνέπειες για όλους. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσει το ότι θα τηρηθούν και θα γίνουν σεβαστές όλες οι θεμελιακές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα πρέπει το κοινωτικό δίκαιο, η ενωμητάξη επίσης να γίνει σεβαστή κατά την εν λόγω διαδικασία. Δεν χρειάζεται σε εσά εδώ να σας τονίσω το ότι η νομική πλευρά των πραγμάτων είναι πολύ σημαντική. Οπότε και όλοι μας θα έχουμε επικοδομητική στάση. Και θέλουμε οι σχετικές συνομιλίες και πραγματεύσεις να γίνονται στα πλαίσια της συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τονίζεται βέβαια το πόσο άρρηκτη είναι η σχέση μεταξύ της πολιτικής διαδικασίας και της νεωματικής πτυχής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτή η περιπλοκότητα είναι αποκοίημα της ένομης τάξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε εδώ κάποια στοιχεία στοιχεία που αφορούν το δίκαιο και θα τα ακούσουμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικά για την ε, διαπραγμάτευση, την αποχώρηση, αλλά και για το μέλλον. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι εμείς οι ευρωβουλευτές έχουμε επίγνωση του ότι οι συνέπειες του Brexit πρόκειται να εμπλέξουν τους Ευρωπαίους και αυτό έχει σχέση με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς σε ποιο συναγματικό, θεσμικό, νομικό πλαίσιο κινούμεθα στο οποίο και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά όλα τα ζητήματα. Οπότε και η σημερινή ακρόαση είναι στα πλαίσια της δουλειάς του Κοινοβουλίου για να προλυάνει το έδαφος και να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Uh, thank you, σε ευχαριστούμε που ήρθες να μας μιλήσεις. Όποτε και αρχίζουμε το πρώτο μέρος της ε, ακρόασης. Και πρώτα-πρώτα θα ακουστεί η φωνή της Σκοτίας. Ο κύριος James Γουλφ, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας, ο, εισαγγελίας αερίου πάγου, ας πούμε, της Σκοτίας. Yeah, 10 minutes or so. Έχετε περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να παραστώ ενώπιον της Επιτροπής σας. Το Brexit θα έχει σημαντικές νομικές συνέπειες για όλους μας. Ε, εγώ ως ε, ανώτατος εισαγγελέα ε, είμαι ο ανώτατος αξιωματούχος νομικός και υπεύθυνο του συστήματος δίωξης στη Σκωτία. Φαντάζεστε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τα θέματα που μπορώ να συζητήσω. Η θέση της κυβέρνησης Σκωτίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή και δημόσια, όπως επίσης και η θέση της σε σχέση με το συνταγματικό μέλλον της Σκωτίας. Όπως γνωρίζετε, το Brexit έχει συνεχίσει να έχει πολιτικές συνέπειες για τη Σκοτία. Ε, θα έχει επίσης ε, συνέπειες για τις μελλοντικές εξουσίες ε, του Κοινοβουλίου της Σκοτίας. Στο, στη σύντομη παρέμβασή μου δεν θα σχολιάσω για τα ζητήματα αυτά, απλώ θα παρουσιάσω κάποιες από τις τεχνικές νομικές συνέπειες του Brexit. Για να μπορέσω λοιπόν ε, να τις θέσω στο σωστό πλαίσιο από ε, απόψεως σκοτίας, πρέπει να πω ορισμένα πράγματα για την, τον χαρακτήρα ε, πολλαπλής δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης και την... Ε, κατανομή των ε, νομοθετικών και εκτελεστικών εξουσιών σε σχέση με τη Σκοτία. Η Σκοτία είναι ένα από τα τρία νομικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει το ε, δικό της ε, σύστημα το νομικό πριν καν από τη δημιουργία του Ηνωμένου Βασιλείου και αντλεί παραδόσεις από τις δύο μεγάλες νομικές παραδόσεις της Ευρώπης. Η Σκοτία έχει πάρα πολλά κοινά ε, στοιχεία με το νομικό σύστημα της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, όμως ε, πολλοί τομεί, όπως η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας, το οικογενειακό δίκαιο και το ποινικό δίκαιο είναι ξεχωριστά. το κεκτημένο βεβαίως είναι τμήμα της νομοθεσίας που ισχύει στη Σκωτία, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι, υπάρχει κάποια νομοθεσία η ε, οποία προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ίδια τη Σκωτία εντό του, του Ηνωμένου ε, Βασιλείου. Ε, υπάρχει ο νόμος Σκωτίας του 1998 που δίνει εκτελεστικές και νομοθετικές αρμοδιότητες μοιρασμένες μεταξύ του Σκοτσέζικου Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης. πολύ σημαντική τομείς όπως η γεωργία και η αλία, το περιβάλλον και η δικαιοσύνη ε, ε, είναι τομείς ο οποίους έχει πολύ σημαντικές αρμοδιότητες σκοτσέζικο ε, κοινοβούλιο ε, συνήθως το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο εξασφαλίζει την έναρξη ισχύω της νομοθεσίας για τα θέματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα. Ε, όμως, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μέσω συμφωνίας, η σχετική νομοθεσία μπορεί να εφαρμόζεται σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται όλος ιδιαιτέρως ε, για τα, τις συνέπειες του Brexit ε, σε σχέση ε, με την νομική συνέχεια του συστήματος. Θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα για τις επιχειρήσεις και η κυβέρνηση Σκοτίας θέλει να εξασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου και την συνέχεια του νομικού συστήματος, όπως επίσης και τη διατήρηση του νομικού καθεστώτος και των πολιτικών της αρμοδιότητός τους. Ε, η κυβέρνηση Σκωτίας ε, θα συνεργαστεί με ε, την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ομοθεσία που θα χρειαστεί στο πλαίσιο του Brexit για να εξασφαλιστεί η νομική συνέχεια και η ασφάλεια δικαίου. Θα ήθελα να σας εξηγήσω κάποια από τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Καταρχάς, πρέπει να ε, δούμε το θέμα της συνοχιζόμενης ισχύω των νόμων που ισχύουν εντός της Σκοτίας. Υπάρχει ένα τμήμα εφαρμοστικού νόμου ε, που λόγω της εγχώριας ισχύω τους θα εξακολουθήσουν να ισχύουν εξαρτήτως Brexit, όμως υπάρχει και ένα τμήμα ενωσιακής νομοθεσίας ε, που προκύπτει από τις συνθήκες και κυρίως προκύπτει από κανονισμούς που ισχύει χωρίς εγχώρια εφαρμοστικά μέτρα στην Σκοτία ε, ε και υπάρχει κάποια νομοθεσία η οποία δυστυχώ θα χαθεί αν δεν γίνει τίποτε για να διατηρηθεί μετά από τον Brexit. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα εξακολουθούν να ισχύουν οι νόμοι αυτοί ε, στο πλαίσιο τη ε, σκοτία μετά την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία θα εξακολουθεί να ισχύει αποτελεσματικά και με σωστό τρόπο. Σε πολλού τομεί μπορεί να ε, γίνει αυτό χωρίς καμία αλλαγή. Σε μερικές περιπτώσεις όμως πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να ισχύει αποτελεσματικά και με το σωστό τρόπο. Κάποιες είναι τεχνικές προσαρμογές, άλλες σημαίνουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές πολιτικής και ο χαρακτήρας και το επίπεδο των επιλογών ε, ποικίλουν. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις επίσης και για, ε, για, τα απαραίτητα, για την απαραίτητη νομοθετική, την κατάλληλη νομοθετική μέθοδο για να γίνουν οι αλλαγές αυτές. Χρειάζεται βέβαια με, μεταξύ των κρατών μελών συνεργασία, ε, γιατί υπάρχουν κάποια, ε, κάποιοι τομεί που δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με μονομερή δραστηριότητα είτε του Ηνωμένου Βασιλείου είτε τη Σκωτία. και αναφέρομαι κυρίως στη συνεργασία για ζητήματα ε, πολιτικής δικαιοσύνης, ε, αμοιβές αναγνώρισης και εφαρμογής των αποφάσεων. Ε, επειδή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των αμοιβαίων διακανονισμών για ζητήματα ποινική δικαιοσύνης και σχετικής συνεργασίας, έχω αναφερθεί πολλές φορές στη σημασία διατήρησης αυτών των διακανονισμών για να μπορέσουμε να καταπολεμούμε το έγκλημα. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι εύκολο να τα αναφέρει κανεί σε γενικό επίπεδο. Το να μπορέσουμε όμω στην πράξη να τα λύσουμε σημαίνει ε, ότι χρειάζεται λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων νομικών καθεστώτων. Η ε, κυβέρνηση της Σκωτία έχει αναφέρει ότι ανεξαρτήτως των όρων Brexit ε, η συνταγματική θέση της Σκοτίας ε, θα αλλάξει ε, για τους λόγους που εξήγησα. Υπάρχουν και κάποια ε, τεχνικά νομικά ζητήματα τα οποία εμείς στη Σκωτία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την νομική συνέχεια και την ασφάλεια δικαίου. Εν ολίγη στην ακαιρεότητα, την συνεχιζόμενη ακαιρεότητα της εσωτερικής μας ένομης τάξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε τον δεύτερο ομιλητή, τον ε, Έτεν Τάναμ από το Trinity College του Δουβλίνου. Έχετε το λόγο. Α, συγγνώμη, κυρία Έτεμ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω δεν είμαι νομικός, ε, είμαι ειδική στον τομέα των πολιτικών επιστημών και θα μιλήσω για τις επιπτώσεις ε, του Brexit για την περιοχή της Ιρλανδίας, της ε, Βόρειας Ιρλανδίας και την περιοχή την διασυνοριακή. Βεβαίως έχει αμφισβητηθεί, όπως ξέρετε, το σύνορο μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας και η Συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής το 1998 σταμάτησε τη βία, βοήθησε να υπάρξει κατανομή των αρμοδιοτήτων και μια συνεργασία η οποία βεβαίως ε, έγινε πιο έντονη μέσω της χρηματοδότησης ε, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Η συμφωνία λοιπόν της Μεγάλης Παρασκευής έχει αμφισβητηθεί μετά από το δημοψήφισμα για το Brexit. 55,8 των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας ψήφισε υπέρ της παραμονής και 85% των καθολικών. Όπως ξέρετε επίσης, ακόμα και η Sinn Féin έκανε έκκληση για την παραμονή πριν από το δημοψήφισμα. Η συνεργασία στην περιοχή των συνόρων είναι κάτι που σαφώς σταθεροποιεί την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 30.000 άτομα κάθε μέρα περνάνε τα σύνορα, 1,8 εκατομμύρια τον μήνα. Πρόκειται για ένα σύνορο 500 χιλιόμετρων με μικρές ε, κοινότητες υπάρχουν περίπου 300 διαφορετικά σημεία περάσματα. Είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει έλεγχος. Όσον αφορά το εμπόριο για το 2015, τα στοιχεία που έχουμε είναι 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικές εξαγωγές λοιπόν της Ιρλανδίας ε, προς την Βόρεια Ιρλανδία. οι ε, τοπικές εμπορικές συναλλαγές είναι κάτι που θα συνεχιστούν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα από την Ιρλανδία στη Βόρεια Ιρλανδία. Μεγάλη αβεβαιότητα επικρατεί σήμερα όσον αφορά τι διαπραγματεύσει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανεί δεν ξέρει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανεί προβλέψει όσον αφορά το ε, αποτέλεσμα και τι επιπτώσει για την ε, πολιτική τη Ιρλανδία. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε απολύτω κανένα σχεδιασμό σήμερα. Το 1942 η κοινή ε, περιοχή που έχει καθοριστεί μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας με συγκεκριμένες διευθετήσεις ε, θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Δεν καλύπτονται όμως εδώ όλοι οι τομείς του ελεύθερου εμπορίου και των ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα σενάρια για την διευθέτηση αυτών των εμπορικών συναλλαγών μετά το Brexit, ηλεκτρονική έλεγχη, σηματοδότηση, καταχώρηση των οχημάτων. Υπάρχουν όμως και άλλου είδους σενάρια, όπως παραδείγματος χάρη να ελέγχονται μόνο κάποια δειγματοληπτικά οχήματα έτσι ώστε να δείξουμε ότι δεν θέλουμε να υπάρξει ένα πραγματικά σκληρό, όπως θα το λέγαμε, σύνορο, κλειστό σύνορο. Άλλα σενάρια, κάποιες ε, διευθετήσεις για κάποιους συγκεκριμένους τομείς, βάσει των ε, σημαντικών τομέων για την οικονομία βάσει της ε, Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, αγροδιατροφικά προϊόντα, να υπάρχουν δηλαδή κάποια τελωνία, αλλά όχι στα σύνορα, αλλά 10 με 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα, για να μην επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση που επικρατούσε πριν την προσχώρηση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα σενάρια για τη συνεργασία η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει στην Τελωνιακή Ένωση ακόμα και αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει πλέον σε αυτήν. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Κάποια από αυτά τα σενάρια που παρουσιάσαμε είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικά. Σαφώς θα πρέπει να προβλεφθούν τρόποι διευκόλυνσης και απλοποίησης, ιδιαίτερα αν αποφασιστεί να υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι. Η θέση του Σινφέιν είναι σαφής, βαθιά ιδεολογική αντίθεση για ένα κλειστό σύνορο με αυστηρούς ελέγχους, κάτι βεβαίως που είναι τελείως διαφορετικό ε, όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία και το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων πολιτική βούληση και διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα, όπως σας είπα, ποιο θα είναι το τελικό σενάριο που θα επικρατήσει. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική διαπραγμάτευση με οικονομική στήριξη και βεβαίως η στήριξη από μέρους της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Ιρλανδίας θα είναι καθοριστική ε, για οποιοδήποτε σενάριο επιτευχθεί και επιλεγεί. Όσον αφορά την Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, η οποία βεβαίως δίνει μεγάλη έμφαση στη συνεργασία και στη μη ύπαρξη ενός αυστηρά κλειστού συνόρου. Από τη στιγμή που μέσω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης άρχισε να ισχύει το ειδικό πρόγραμμα για την διαθέτηση των συνοριακών ε, ανταλλαγών και των εμπορικών ανταλλαγών. Αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντικατασταθεί, να διευθετηθεί από τις νέες αποφάσεις. Το θέμα τώρα της υπηκότητας. Βάσει της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν την Ιρλανδική, την Βρετανική ε, ή και τις δύο υπηκότητες. Το άρθρο 11 της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει αναθεώρηση και τροπολογία. Αυτό μάλιστα έγινε το 2006. Είναι η λεγόμενη συμφωνία του Αγίου Ανδρέα, St. Andrews Agreement. Η λειτουργία λοιπόν του αρμόδιου οργάνου για τις διασυνοριακές εμπορικές ε, ανταλλαγές και τη συνεργασία είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευθετηθεί βάσει των νέων διατάξεων που θα ισχύουν μετά το Brexit. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση λοιπόν να επανεξετάσουμε τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και να αναγνωριστούν οι τελικές διαθετήσεις το 2015 μόνο μια μικρή πλειοψηφία, περίπου το 32% των καθολικών ήθελαν επανένωση ε, της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία και μόνο 14% του συνολικού πληθυσμού υποστήριζε κάτι τέτοιο, πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά το Brexit. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι η Βόρειος Ιρλανδία και η Ιρλανδία θα επηρεαστούν με μοναδικό τρόπο αρνητικά από το Brexit. Η κακή διευθέτηση του θέματος ε, της ε, περιοχής των συνόρων είναι κάτι που σε αυτός μπορεί να έχει πολύ σοβαρότερες αρνητικές επιπτώσεις για όλη την περιοχή. Το θέμα της ταυτότητας θα πρέπει να διευθετηθεί με μια λεγόμενη ευέλικτη λύση. Αυτό εξάλλου ε, αποτελεί και τμήμα του πρώτου πορίσματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Brexit. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε λίγα λεπτά για να συζητήσουμε αυτές τις δύο πρώτες ε, παρουσιάσεις και ομιλίες. Δεν θέλω εγώ να κάνω την πρώτη ερώτηση στον πρώτο ομιλητή. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, στο Scottish Act του... Ναι, under the devolved competencies must be ε, compatible with EU law.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 Και σαφώς και το Βρετανικό, η Βρετανική κυβέρνηση ενδεχομένως ε, θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο της Σκοτίας να αυξήσει τις ε, αρμοδιότητες και τις εξουσίες του. Εάν δεν υπάρξουν ε, αλλαγές στον τομέα αυτό, και όπως διαβάζουμε το σημείο 10 του αντίστοιχου εγγράφου με κατευθυντήριες γραμμές όπως έχει δημοσιευθεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυρία Νίτλερ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση στον πρώτο ομιλητή μας δείξατε ότι υπάρχουν ξεχωριστές αρμοδιότητες για τη σκοτία στην ομιλία σας. Όταν ολοκληρωθεί το Brexit, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίζει να πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο εφόσον έχει ενσωματωθεί στην νομοθεσία σας. Εδώ είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον δεν θα ανήκει στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι θα γίνει με τα δικαστήρια της Σκοτίας, τι θα γίνει στην πράξη και τι θα γίνει βάσει των ε, ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας στη Σκοτία. Έχω και μία ερώτηση προς την δεύτερη ομιλήτρια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του hard και του soft border, όπως είπατε, ενώ δηλαδή συνόρου κλειστού με αυστηρούς ελέγχους και μιας πιο ευέλικτης κατάστασης. Καταλαβαίνω ότι οι αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της περιοχής αυτής μπορεί να είναι τεράστιες, καταστροφικές. Δεν καταλαβαίνω όμως ακριβώς ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτών ε, συνόρων. Φαντάζομαι ότι η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει λίγο τα πράγματα, να αποφευχθεί η γραφειοκρατία. Αλλά εξηγήστε μου, με το πέρασμα ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων καθημερινά, όπως μας είπατε, πώς θα ρυθμιστούν αυτά τα προβλήματα και ποια είναι πραγματικά η διαφορά μεταξύ του soft και του hard border. Για να απαντήσω πρώτα αυτά που εμένα ρωτήσατε και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Αυτό που βασικά ήθελα <clears throat> να αναδείξω με την ομιλία μου είναι το ότι έχει κάποιες αρμοδιότητες, κάποιες ευθύνες η Σκωτία για διάφορες πολιτικές που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οπότε η κυβέρνησή μας και το κοινοβούλιο μας θα έχουν τη σχετική ευθύνη με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα έχουμε την ευθύνη ούτω ώστε να υπάρξει συνέχεια στο δίκαιο και ασφάλεια δικαίου. Και σε συνεννόηση με την Βρετανική κυβέρνηση θα τα εξασφαλίσουμε όλα τούτα. Για τα σχετικά πρόκειται να νομοθετήσει η Βρετανία. Δεν μπορώ να σας πω τώρα περισσότερο. Τώρα, αυτά που αφορούν το δικαστήριο που με ρωτήσατε και κάποιες τεχνικές ερωτήσεις για τεχνικά ζητήματα που επισήμανα. Ε, βέβαια και η νομολογία του δικαστηρίου θα συνεχίσει να έχει σημασία για διάφορου τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου που επηρεάζουν την ε, Εθνική Ένωμη Τάξη. Θα ήταν πρόημο να πω οτιδήποτε σχετικά. Ε, βέβαια και έχουμε κάποια ουσιαστικά θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σύντο χρόνο θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά που θα αναδυθούν. Γι' αυτό είπατε για το soft σύνορο. Αυτό είχε σήμερα, δηλαδή κανείς διασχίζει τα σύνορα, πάει από την ε, Ιρλανδία στη Βόρεια Ιρλανδία, πήγε και ο κύριος Μπαρνιέ πρόσφατα και εκτός από τις αλλαγές ε, ε, στη σηματοδότηση του δρόμου δεν καταλαβαίνει κανείς ε, το ότι διέβη τα σύνορα. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί. Και αν δεν υπάρχει ελευθερία διακίνησης και ταξιδίου, θα είχαμε hard σύνορα, σκληρά, ε, και αυτό θα ήταν καταστροφικό. Έχουμε τώρα ε, δάσκαλους, ε, διάφορους που κάνουν δουλειές και διαβαίνουν τα σύνορα συνέχεια. Αλλά πάντως δεν το θέμα δεν είναι μόνο το ζήτημα του να ε, σύνορα για να δουλέψει, αλλά και για να αναζητήσει κάποιες υπηρεσίες. Να, ας πούμε ακόμα και νοσοκομιακά δρούν διασυνοριακά. Έχουμε αστυνομικά θέματα και εκεί. Εμείς φυσικά και θέλουμε, όπως και έχει ενδιαφερθεί να το φροντίσει και η Πρωθυπουργός με το καθεστώς που ισχύει σήμερα. Τώρα, για το εμπόριο θα πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε τα αρνητικά όσον αφορά τους περιορισμούς του ελευθερίου εμπορίου. Να έχουμε ενιαία αγορά σε όλο το νησί. Ιδάλλως θέλουμε να περιοριστούν τα αρνητικά αποτελέσματα κάποιων σκληρών σύνορων που θα είναι πολύ καταστροφικά για τις εταιρείες. 100 ευρώ κάθε μέρα θα κοστίζουν αυτά τα σύνορα. Λόγω γραφειοκρατίας. Τόσο θα κοστίζουν στις εκκλησίες, στις εταιρείες. Αυτό το παρτισσόκο σύστημα ελέγχου των ε, εμπορευμάτων που διασύζουν τα σύνορα. Καταστροφικό θα ήταν οικονομικά αυτό και για τις μικρές εταιρείες αλλά και για τις μικρές εκμεταλλεύσεις και ε, εταιρείες για γεωργικά προϊόντα. Οπότε θα επηρεαστεί και το εμπόριο και η ζωή γενικά των ανθρώπων. Τον υπάρχουν τέτοια σκληρά σύνορα. Υπάρχουν γίνει κάτι προτάσεις για ηλεκτρονική ετικετοθεσία, ε, διάφορες λύσεις, αν δεν γίνεται τίποτα άλλο με τα σύνορα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος, κυρία Μπερζερό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την Ιρλανδία εκπρόσωπο είναι η ερώτησή μου. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι εξίσου καλά δομημένη με τη Σκοτία από απόψεως θεσμικής και υπάρχουν εκπρόσωποι της Βόρειας Ιρλανδίας που μπορούν πραγματικά να εκφράσουν με σθένος την άποψη των Βόρειο Ιρλανδών σε σχέση με την ε, βούλησή τους να παραμείνουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τέτοιου είδους δομές όπως στη Σκοτία. Αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Ε, καταρχάς, ε, τα πολιτικά κόμματα ε, στην Βόρεια Ιρλανδία είναι κατά του σκληρού συνόρου. Επίσης υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιρλανδία γιατί η εκτελεστική εξουσία έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αλλά υπάρχει ε, μια κυβέρνηση υπό την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ε, και ε, ούτως ή άλλως η κατάσταση ως προς αυτό είναι ίδια με τη Σουαλία και τη, Σκωτία. και τη, και επειδή κατέρευσε η εκτελεστική εξουσία μετά έγιναν εκλογές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε προεκλογική εκστρατεία αυτή τη στιγμή μετά νομίζω ότι θα μπορέσουν περισσότερο να συνεργαστούν επί του ναι. ζητήματος Brexit τα διάφορα διάφορα πολιτικά κόμματα. Όμως για την ώρα ε, οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ ε, του ε, Sinn Féin και των άλλων πολιτικών ομάδων, των πάλι πολιτικών κομμάτων για το Brexit, ο Brexit όπως γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα, είναι ότι επικεντρώνονται κυρίως στην στην προσπάθεια αποφυγής ενός σκληρού, ενός hard border. Το ερώτημά μου είναι προς τον ε, εισαγγελέα Ριού Πάχου της Σκοτίας. Ε, αναφερθήκατε στο νόμο για τη Σκοτία. Αν κατάλαβα καλά, και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπάρχει το χειρότερο πιθανό σενάριο, δεδομένου δεδομένης της κυρίαρχης πολιτικής ε, του Westminster, τι θα γίνει με τις εξουσίες που έχει η Σκοτία. Υπάρχουν πραγματικές εξουσίες ε, που δεν μπορούν να τις καταργήσουν στο Westminster. Σας ερωτώ, γιατί αν κατάλαβα καλά, ε, το Κοινοβούλιο της Σκοτίας ε, είναι... Είναι, είναι, μια, είναι, μια, είναι, η κυριαρχία είναι κυριαρχία ε, της Σκοτίας, ενώ του Westminster είναι κοινοβουλευτική ε, η ε, κυριαρχία. Ναι, να προσπαθήσω να σας απαντήσω. Πηγαίνουμε πίσω στα θεμέλια της δημιουργίας του Ηνωμένου ε, Βασιλείου. Ε, κάποια πράγματα είναι γραμμένα στο Σύνταγμα της Σκοτίας και από εκεί προκύπτει το νομικό σύστημα ε, βάσει του οποίου προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να εξασφαλίζουμε το γεγονός ότι η ένομη τάξη της Σκοτίας διατηρείται ε, μετά την ένωση ε, του 1707 ε, υπήρξε ένα, ένας νόμος, αυτός ο νόμος για τη Σκοτία του 1988 η οποία καθιστά σαφές ότι το Κοινοβούλιο της Σκοτίας είναι ένα μόνιμο τμήμα της συνταγματικής δομής του Ηνωμένου Βασιλείου και εγώ δεν θεωρώ ε, ότι υπάρχει το σενάριο που αναφέρατε εσείς. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δεν θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό αυτό το οποίο είπατε. Okay. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Ντανούτα. Ναι, θα ήθελα να καταλάβω το εξής ε, τον ε, εισαγγελέα ε, του Αρίου Πάγου της Σκοτίας. Το ερώτημά μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Ε, αυτός ο μεγάλος, αυτό το μεγάλο, ε, μεγάλος νόμος ανάκλησης πώς θα καλύψει όλο αυτό το θέμα των αρμοδιοτήτων γιατί είπατε ότι υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες του Σκοτσέζικου Κοινοβουλίου επί συγκεκριμένων τομέων και για άλλους τομείς όχι. Τι θα κάνει λοιπόν το νόμο σχετικά με αυτό το θέμα και είπατε στην αρχή ότι η θέση της κυβέρνησης της Σκοτίας είναι θέμα δημόσιο. Ε, και το ερώτημά μου είναι το εξή. Στο πλαίσιο εκχώρησης εξουσιών με, το, με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ποιο βαθμό η διαφάνεια στη διαδικασία λήψη αποφάσεων που επηρεάζει και τη Σκωτία εμέσως, σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτό το στοιχείο, υπάρχει καθόλου αυτό το στοιχείο, υπάρχει δηλαδή κάποια νομική δέσμευση, κάποια δέσμευση μέσω συμφωνία από πλευρά Βρετανική κυβέρνηση να είναι διαφανή σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία του Brexit. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για το πρώτο σας ερώτημα που έχει να κάνει με τον νόμο περί ανάκλησης. Ε, η Βρετανική κυβέρνηση και η Λευκή της Βίβλος αναφέρει ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα, τις διάφορες εκχωρημένες εξουσίες ε, στα διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως δεν έχουμε δει ακόμη το ε, νόμο αυτό, οπότε ε, νομίζω ότι θα καταλάβετε αν δεν σχολιάσω περαιτέρω η κυβέρνηση της Σκοτίας ε, βεβαίως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, για τις διατάξεις αυτές ε, του νόμου και θα συνεργαστεί, θα συζητήσει με τη Βρετανική κυβέρνηση κατά σε σχέση με το κατά πόσο καλύπτει ο νόμος αυτός τις διάφορες ανησυχίες μας. μου θέσατε ένα ερώτημα για τη διαφάνεια. Δεν... Ε, ε, δεν θέλω να δείξω ε, έλλειψη σεβασμού, αλλά δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά τι, που εστιάζουμε αυτή τη στιγμή. πολύ συχνά εμείς υποβάλλουμε εκθέσεις σε σχέση με τις εξελίξεις από πλευρά Σκοτίας για το Brexit. δείχνουμε λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι αναφερόμουν περισσότερο στα διάφορα επίπεδα γιατί έχουμε ακούσει από ε, αξιωματούχους της κυβέρνησης της Σκοτίας σχόλια που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι κάποια έγγραφα που έχουν να κάνουν με το Brexit ε, δεν είναι γνωστά ε, στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Σκοτίας πριν ε, κυκλοφορήσουν στις Βρυξέλλες και αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει κάποια διαφορά επίπεδου ε, ναι, αυτά δεν είναι, τεχνικ... δεν είναι νομικά ζητήματα, ε, είναι η απάντηση. Ε, είναι ζητήματα διαπραγματεύσεων ε, και διαλόγου. Ε, θα είναι καλύτερα και είμαι ε, σίγουρος ότι οι Υπουργοί με πολύ χαρά θα παραστούν στην Επιτροπή σας και σε άλλες Επιτροπές να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, ερωτήματα τα οποία δεν είναι καθαρά τεχνικής φύσεως. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να συνεχίσουμε τώρα με το δεύτερο τμήμα της ε, ακρόασής μας ε, και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα για το αστικό δίκαιο από τον κύριο ε, Χες, που είναι ο Διευθυντής του Ινστιτού Max Planck για το δικονομικό δίκαιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας μιλήσω συνοπτικά για την σημασία του Brexit όσον αφορά τις διασυνοριακές διαφορές στην Ευρώπη. Έχω χωρίσει την εισήγησή μου σε τέσσερα μέρη. Πρώτα-πρώτα να σας πω ποιοι είναι οι τομείς που θα επηρεαστούν. Πρώτα-πρώτα έχουμε τα θέματα οικογενειακού δικαίου. Κατόπιν έχουμε τα θέματα εμπορικού δικαίου ε, αυτά θα αναλυθούν κάπως περισσότερο. Βεβαίω έχουμε οικογένειες που επηρεάζονται και στην Βρετανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα αυτά η αποχώρηση θα τα επηρεάσει. Επίσης να μιλήσουμε για τις ε, συνέπειες του Brexit σε σχέση με την ε, Σύμβαση Υπαρθμών των Βρυξελών γιατί θα πρέπει να δούμε το τι μπορούμε να πετύχουμε μέσω της σύμβασης του Λουγκάνο και τη νομοθεσία ή το νομοθέτημα για την κατάργηση κάποιας νομοθεσίας. Η 29η Μαρτίου του 2019 αυτή είναι η ημερομηνία κλειδί για το τι θα γίνει, τι θα γίνει και τι χρειάζεται να συμφωνηθεί. Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα νομοθετήματα που είναι πρόσφατα. Είναι κάποιοι κανονισμοί που με το Brexit θα καταργηθούν θα σταματήσουν να υπάρχουν όλες αυτές οι νομοθετικές πράξεις. Για να δούμε πρώτα πρώτα τι γίνεται όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο. Εδώ έχουμε δύο βασικά νομοθετήματα. Πρώτα πρώτα την, ε, τον κανονισμό των Βρυξελών που ε, έχει σχέση με διαζύγιο, με γονική μέρημνα, με υποχρεώσεις των γονέων και επίσης με την ε, διασυνοριακή εκτέλεση αποφάσεων. Επίσης έχουμε τον κανονισμό για την διατροφή, πολύ σημαντικός. Στην πράξη έχει πιάσει το από αυτή η νομοθεσία. Επίσης έχουμε και το θέμα των μικροδιαφορών, δηλαδή διαφορές που αντιστοιχούν σε λίγες εκατοντάδες ευρώ. Θα πρέπει να πώς θα εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις διασυνοριακά. Και έχουμε αυτό το όριο του ε, ναι, το, το, το ορόσημο, να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά του κανονισμού οι οποίοι θα καταργηθούν. Τι θα γίνει με τα διαζύγια, τίποτα. Τι θα αντικαταστήσει αυτή την νομοθεσία και όσον αφορά τι διατροφέ, τα πράγματα είναι λίγο πιο ρόδινα. Γιατί έχουμε τη σχετική σύμβαση τη Χάγη που έχει συλλογικό χαρακτήρα, δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσον αφορά σε σχέση μάλλον με τα πιο αποτελεσματικά κοινοτικά το θέμα είναι ότι κάθε φορά πρέπει να θέτουμε δύο ερώτημα. Τι θα γίνει παραδείγματο χάρη με μελλοντικέ ε, διαφορές, διαμάχε μετά το Brexit. Επίσης, τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να ρυθμιστεί μία διαφορά η οποία ξεκίνησε πριν την αποχώρηση, πριν το Brexit και αν μπορούμε να την συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Αν υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι, ποια διάρκεια θα έχουν. Για τις ε, μελλοντικέ διαφορές νομίζω ότι το θέμα είναι πολιτικό και πρέπει να δοθεί πολιτική απάντηση. Τώρα, όταν αφορά κάποιες ε, οικονομικές διαφορές, εμπορικές διαφορές, Βρυξέλλες 1, αυτός είναι ο πρώτος κανονισμός, ο οποίος ε, ισχύει εδώ. Όσον αφορά όμως την ε, συνεργασία και τον κανονισμό που διέπει διαφορές ε, οικονομικές εμπορικές, αυτές πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο, δεν θα ισχύει πλέον αυτός ο κανονισμός και σε κάθε περίπτωση αν ξεκινήσει μια διαδικασία πριν το Brexit θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για το πώς ακριβώς θα συνεχιστεί. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, αποδείξεις ε, όσον αφορά την ισχύ της ε, σύμβασης της Χάγης του 70 του 65 μέχρι τώρα όπως ξέρετε έχει τελείως διαφορετική ε, ισχύ στο ιδιωτικό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο η σύμβαση δηλαδή Ρώμη 1 και Ρώμη 2 οι οποίες κανονικά θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις διαφορές ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως, σε περίπτωση διαφοράς στο εσωτερικό ε, της ε, Μεγάλης Βρετανίας δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν να ισχύουν ναι ή όχι αυτές οι διατάξεις και η σύμβαση που ισχύει σήμερα. Τώρα, ποιες μπορεί να είναι και ποιες θα είναι οι πρακτικές συνέπειες ε, για τις διαφορές ε, και στην Ευρώπη, αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία. Όπως ξέρετε, σήμερα το Λονδίνο συνεχίζει να είναι ένας πολύ μεγάλος, ε, ένα πολύ μεγάλο κέντρο για την επίλυση διαφορών, ιδιαίτερα αστικού δικαίου και αυτό διότι αποτελεί για τις οικονομικές, χρηματοπιστωτικές διαφορές, διαφορές που αφορούν το ναυτικό δίκαιο και βεβαίως πολλές φορές επιλέγεται και από ζευγάρια με οικονομική άνεση το Λονδίνο για την επίλυση των διαφορών του σε θέματα διαζυγίου το θέμα παραδείγματο χάρη του πτωχε... Ε, των πτωχεύσεων, το πτωχευτικό δίκαιο επίσης, ε, πολλές φορές ε, εφαρμόζεται και επιλέγεται το Λονδίνο για την εφαρμογή των αποφάσεων. Γιατί το Λονδίνο είναι τόσο πολύ σημαντικός προορισμός για αυτού του είδους της ε, αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα για τη γλώσσα, γιατί η αγγλική γλώσσα είναι η διεθνής γλώσσα για την επίλυση εμπορικών διαφορών. Με εξειδικευμένους λοιπόν δικαστές, το διαδικαστικό δίκαιο στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και με αυτόν τον τρόπο μπορεί οι διαδικασίες να είναι αποτελεσματικές, ταχείες. Γι' αυτό και επιλέγεται το Λονδίνο. Υπάρχουν όμως δύο σημεία, τα οποία τα έχω εδώ σημειώσει με κόκκινο χρώμα, το ένα είναι ότι το αγγλικό δίκαιο, το βρετανικό δίκαιο, έχει ένα πόδι, αν θέλετε, στο κοινοτικό δίκαιο και δεύτερον το θέμα των αποφάσεων του ενός αγγλικού δικαστηρίου που ε, αυτομάτως ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν κοιτάξετε τον ιστότοπο του ε, αντίστοιχου commercial law δικαστηρίου του Λονδίνου βλέπετε όλες αυτές τις πιθανές ε, διευθετήσεις μιας απόφασης που λαμβάνεται από ένα αγγλικό δικαστήριο στο Λονδίνο και τις δυνατότητες ε, που υπάρξουν συνύπαρξης με το κοινοτικό δίκαιο. 500 τουλάχιστον διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου, εκ των οποίων το 80%, το 80% αυτών, ε, ένα από τα δύο μέρη δεν είναι Βρετανός υπήκος ή Βρετανική εταιρεία. Αυτό είναι μια μοναδική, μοναδική περίπτωση παγκοσμίως. Το 60% αυτών των διαφορών αφορούν ποσά που ξεπερνούν τις 300.000 λίρες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει και την σημασία αυτών των διαφορών από οικονομικής απόψεως. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες της γερμανικής επικράτειας. Μπορείτε να το διαβάσετε και πολύ σύντομα θα περάσω στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές ε, τις καταστάσεις που θα προκύψουν ε, μετά την ε, αποχώρηση, τι θα γίνει όταν πάψει να ισχύει η Σύμφωση Βρυξέλλες 1 και πολύ συγκεκριμένα η Σύμβαση των Βρυξελών του 68 μπορεί να αντικαταστήσει την ε, Σύμβαση Βρυξέλλες 1. Πρόκειται για μια διεθνή σύμβαση βεβαίως, η οποία όμως κατά την άποψή μου ανήκει στο κοινοτικό δίκαιο, στο κοινοτικό εκτιμένο Πρόκειται λοιπόν για ένα τμήμα αναπόσπαστο του κοινοτικού δικαίου. Δεν είναι λοιπόν λύση αυτή η Σύμβαση των Βρυξελών. Και με αυτόν τον τρόπο επανερχόμαστε στις διμερείς συμβάσεις που ήταν κάτι που ίσχυε από την δεκαετία του 30, διμερείς συμβάσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και κρατών μεμονωμένων. Υπάρχουν έξι τέτοιες συμβάσεις. Εάν κάποιος θέλει να ξαναμπεί σε αυτήν την διαδικασία των διμερών συμβάσεων, διπλασιάζει και τις διαδικασίες αλλά και την αναγνώριση των αποφάσεων. Βλέπετε ότι εδώ λοιπόν θα υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική αρνητική συνέπεια μετά το Brexit. Τι μπορεί κανείς να κάνει. Πολύ σύντομα, είτε κύρωση σύμφασης και συμφωνίας που να διέπει τις διαφορές αυτή και την επίλυση αυτών των διαφορών μετά το Brexit, Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να αποφασίσει να μην ε, ισχύει πλέον το διαδικαστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλη αστάθεια, καθότι μια τέτοια επιλογή, δηλαδή να μην εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση, θα θα υπογραμμίσει μόνο κάποιες από τις πτυχές αυτού του δικαίου. Η σύμβαση του Λουγκάνο, παραδείγματος χάριν, ε, έχει άμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο, πώς θα αντιδράσουν τα άλλα κράτη-μέλη μετά την αποχώρηση του Μεγάλου Βρετανίου. Βλέπουμε, παραδείγματο χάρη, στις, κάτω χώρε, στη Γαλλία και στη Γερμανία υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίε για να εγκαθιδρυθούν σύγχρονες διαδικασίες στην ε, αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε κάποιες από τις διαφορές που μέχρι τώρα ε, είχε προσελκύσει το Λονδίνο να μπορέσουν να μεταφερθούν και να επιληθούν σε κάποιες άλλες πρωτεύουσε. Δεν ξέρουμε βεβαίως ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Καθοριστικό είναι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου να υπάρξει ασφάλεια. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εμπορικές διαφορές υπάρχει ανάγκη, απόλυτη ανάγκη μιας νέας παράλληλης ε, λύσης, παράλληλης αυτής που δίνεται σήμερα βάση του ε, της Σύμβασης Βρυξέλλες 1. Θα πρέπει δηλαδή με έναν ήπιο και ομαλό τρόπο να γίνει μετάβαση από το Λονδίνο σε κάποιους άλλους τόπους όπου θα επιλύονται αυτές οι διαφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε καθηγητά. Τώρα η επόμενη και ο καθηγητής Ντάνκαν Μάχης θα μας τα παρουσιάσει, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κούνη Μέρη του Λονδίνου. Ευχαριστώ. Το σύστημα των ευρεσιτεχνιών είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ε, καινοτομία και για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Από το 1973 έχουμε τη σχετική σύμβαση για την Ευρώπη που ε, με βάση αυτή ε, συγκροτήθηκε το, η υπηρεσία για τις ε, ευρεσιτεχνίες και ε, έχουν προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση 38 κρατη Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ο ετών μπορεί στη συνέχεια να κατοχυρώσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την εφευρεσή του, ας πούμε, σε τουλάχιστον 38 κρατημέλη. Συγγνώμη γιατί με τι τα μπέρδεψα κάπως. Τον Δεκέμβριο του 2012 αποφάσισαν τα κράτη-μέλη ε, με βάση την αναβαθμισμένη συνεργασία να θεσπίσουν διακονισμούς όσον αφορά την συγκρότηση της ενιαίας διαδικασίας κατοχήρωσης ευρεσιτεχνιών. Γιατί αντί να υπάρχουν οι χρεώσεις και τα τέλη χωριστά σε κάθε χώρα μέλος και να υπάρχουν αντίστοιχε διαφορές χωριστά, να υπάρξει ενιαία ευρεσιτεχνία και να συμμετέχουν σε αυτή την ρύθμιση όλα τα μέλη. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, Ισπανία, Πολωνία και Κροατία είπαν ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο σύστημα. Ε, με βάση την αναβασμένη συνεργασία, την ενισχυμένη συνεργασία τέλο πάντων, επίση το 2012 είχαμε την διεθνή συνθήκη που αφορά το ενιαίο δικαστήριο επίλυση των σχετικών διαφόρων. Οπότε έχουμε τώρα και το κατευθυνόμενη διαδικασία όσον αφορά αυτέ τι διαφορέ για την ισχύ των ε, ευρεσιτεχνιών ή για ε, τις παρανομίες ε, τις σχετικές με τις ευρεσιτεχνίες όπως έχουν σήμερα τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό διότι αυτή η συμφωνία για τις ευρεσιτεχνίες απαιτεί τουλάχιστον 13 κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων των τριών κρατών μελών με τις περισσότερες ευρωστεχνίες, δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία. Θα πρέπει αυτές οι τρεις χώρε να έχουν κυρώσει αυτή τη συμφωνία πριν αυτή τεθεί σε ισχύ. Έχει δηλώσει τον Νοέμβριο του 2016 στο Συμβούλιο Εντονιστικότητας του Ηνωμένου Βασίλειο ότι πρόκειται να κυρώσει αυτή την συνθήκη. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται εν αναμονή. επομένω. Και μόλις γίνει αυτή η κύρωση, τότε το ενιαίο δικαστήριο πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί. Είπε τον Βασίλειο ότι βρίσκεται καθοδόν προς την κύρωση και έτσι θα μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία του το σχετικό δικαστήριο. Και όταν αυτό συμβεί θα είναι επίσης εφικτό να τεθούν σε ισχύ σχετικοί κανονισμοί. Άρα κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η έναξη λειτουργία του δικαστήριου. Και όπω σα είπα, ο σχετικό κανονισμό προβλέπει ότι θα προβλέπονται οι ευρεσιτεχνίε σε όλα τα κρατημέλη που έχουν υπογράψει Και το τέλο θα είναι ενιαίο για όλε. Το θέμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο αν θα μπορεί να συμμετάσχει ε, σε αυτόν τον κανονισμό μετά την αποχώρηση, τον Brexit. Σαφώς όχι, αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα στην διαφάνεια αναφέρεται στον κανονισμό ότι αφορά μια ειδική ρύθμιση που αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και έχουμε το άρθρο 142 αυτή της σύμβασης που επίσης ε, αναφέρει τον όρο ειδική ρύθμιση. Άρα η υπηρεσία ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να προβλέψει δικό καθεστώ για το Μέλλον Βασίλειο, τόσο ώστε η χώρα να μπορεί να συμμετάσχει στη σχετική συμφωνία. Και όσον αφορά τον κανονισμό επίση, ε, για να υπάρχει και εκεί αυτή η νέα πρόβλεψη έγκριση ευρεσιτεχνιών. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτή η νέα συμφωνία για τι Ε, είναι μια διεθνή συνθήκη. Επομένω, ισχύουν οι κανόνε. Τη σύμβαση τη Βιέννη για τις συνθήκε. Συνθήκες. Ε, άρα ισχύουν αυτά εκτός εάν υπάρχουν κάποιες διατάξεις κάποιου είδους εξαίρεση. Ρήτρα εξαίρεση, ούτω ώστε να προβλέπεται ότι αν κάποιο μέλο μπορεί να αποχωρήσει. Η ενιαία συμφωνία δεν έχει όμως τέτοια ρήτρα και άρα τα τη σύμβασης της ε, Βιέννης για το δίκαιο των συμβάσεων ισχύουν προκειμένου επίση θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούται να εγκρίνει τώρα αυτήν την ε, συμφωνία. Λόγω του άρθρου 18 της Σύμβασης της Βιέννης, κανείς που έχει προσπόραψει η Διεθνή Συμφωνία δεν μπορεί να ενεργήσει κατά των σκοπών και στόχων αυτής της σύμβασης. Ε, άρα θα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία κύρωσης το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα. Παρ' όλα αυτά η Σύμβαση της Βιέννης λέει στο άρθρο 62 ότι υπάρχει η περίπτωση κάποιας ε, εκβάθρων αλλαγή των ε, συνθήκων που δεν προβλεπόταν. Οπότε τότε θα μπορούσε κάποιο κράτος μέλος να αποσυρθεί από μια διεθνή συνθήκη. Και σε διάφορα σημεία η ενιαία συνθήκη της λέει ότι όλοι οι συμβαλόμενοι ε, πρέπει να είναι κράτη-μέλη. Οπότε, αν αποχωρήσει από την Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε θα έχουμε μια άρδιν αλλαγή συνθήκων που δεν έχει προβλεφθεί και άρα θα είναι προβληματική η λειτουργία αυτής της συμφωνίας εάν παραμείνει ε, στην συμφωνία αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή την ενιαία συμφωνία μετά από τον Brexit. Επ' αυτού έχει νομολογήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την γνωμοδότηση 1 κάθος του 9 και εκεί αναφέρεται σε αυτή τη συμφωνία. Σε αυτή την γνωμοδότηση ορίζει το δικαστήριο ότι έχουμε αυτή τη συμφωνία που αποτελεί, που λέει ότι αυτή η συμφωνία τέλος πάντων ε, ότι αντιβαίνει στο κοινωτικό δίκαιο αυτή η συμφωνία γιατί έχει κράτη-μέλη και μη κράτη-μέλη. Οπότε είπαμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν αναλύσουμε την γνωμοδότηση θα διαπιστώσουμε ότι η πρώτη εκδοχή της συμφωνίας ε, θα αφαιρούσε αρμοδιότητες από τα εθνικά δικαστήρια όσον αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Και αντίστοιχα θα μπορούσε να κάνει τίποτα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και επομένω έχουμε αυτή την γνωμοδότηση που αποστερεί αρμοδιότητες από κράτη-μέλη, επομένως δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν όλες αυτές οι διατάξεις. Τώρα τι έγινε μετά τη γνωμοδότηση. Είχαμε την καινούργια διατύπωση της συμφωνίας για να λάβει υπόψη το ότι έχει προτεραιότητα το κοινοτικό δίκαιο και να καλυφθεί η δυνατότητα της αξίωσης αποζημιώσεων για ε, την παραβίαση του κοινωτικού δικαίου από πλευράς του δικαστηρίου και έτσι με κάποιες προδικαστικές παραπομπές του δικαστήριο να δοθεί μια λύση. Επομένως, μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να συμμετέχει στην Συμφωνία για τις ευρωτεχνίες όπως σας εξήγησα η γνωμοδότηση ένα κάθετος ε, εννέα δεν αποκλείει το να συμμετάσχουν κάποια μη κράτη-μέλη στην νέα συμφωνία. Και το ενιαίο σύστημα ευρεσιτεχνιών είναι συμβατό με την ε, συνθήκη και τη συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως απαιτείται το δικαστήριο να ελέγχει το κατά πόσο τηρείται το διεθνέ δίκαιο. Όμως πρόκειται για διεθνέ δικαστήριο και οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία στο Λονδίνο και άρα θα μπορεί το Ηνωμένο να συμμετάσχει στη συνθήκη διότι το δικαστήριο το σχετικό και όχι τα κράτη-μέλη ε, καλούνται να συμμορφωθούν προς το κοινοτικό δίκαιο. σχετικά αυτά τα λέει το άρθρο 21 του, της Συμφωνίας για τις τεχνίες. Οπότε, αν θα μπορούσε να παραμείνει μέλος της ε, Σύμβασης για τις τεχνίες του Βασίλεια, τότε ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταβολές. Όπως σας ε, είπα, αναφέρεται ρητός ότι τα ε, συμβαλόμενοι είναι τα κράτη-μέλη, άρα θα πρέπει να αναφέρονται συμβαλόμενα κράτη ε, και κάποια κράτη από αυτά τα συμβαλόμενα δηλαδή θα μπορούν να μην είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα γίνουν όμως οι τροποποίησεις της συνθήκες. Έχουμε το άρθρο 87 της Σύμβασης για το Δικαστήριο των και λέει ότι θα μπορούσε το Δικαστήριο να ε, ε, τροποποιήσει την συνθήκη όπου χρειάζεται. Όμως από πολιτικής πλευράς αυτό θα ήταν απαράδεκτο. Και ανταυτού χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διευκρινίσει και να ερμηνεύσει την γνωμοδότηση 1 κάθετος 09 και το, τι ισχύει για να συμμετάσχει στο Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών κάποιο μη κράτος μέλος. Αυτά σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και... Τώρα, η τελευταία ομιλία αφορά το καταστατικό των υπαλλήλων. Ο κύριος Στεφάνου Ροντριγκές ε, θα μας μιλήσει από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Έχετε 10 λεπτά, κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να παραστώ στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις ε, για να ε, σας εξηγήσω το πλαίσιο της παρέμβασής μου. Το ερώτημα ετέθη όσον αφορά το καθεστώς των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, το Brexit, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο επί των κειμένων ε, των σχετικών κανονισμών και που αναφέρονται εδώ στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Ε, δεν θα υπάρξει λοιπόν καμία επανάσταση ε, κειμένων ε, που διέπουν το καθεστώς των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ένωσης. Αντιθέτως, θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό το αντίκτυπο για το προσωπικό βρετανικής υπηκότητας. Ε, θα το εξετάσουμε αυτό σε μία πρώτη φάση, αλλά δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίσουμε και τον αντίκτυπο σε άλλους υπαλλήλου και λοιπό προσωπικό που θα μπορούσε να συνδέεται με το Brexit. Αυτό θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Πρώτη ε, πτυχή άμεσος αντίκτυπος ε, επί των υπαλλήλων και του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρετανών. Να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία για να έχετε μια ιδέα ε, του προσωπικού περί του οποίου πρόκειται πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των ενεργεία υπαλλήλων και προσωπικού και των υπαλλήλων ή προσωπικού ε, που έχουν συνταξιοδοτηθεί. 1.650 άτομα είναι περίπου ε, το προσωπικό εν ενεργεία Βρετανικής υπηκότητας. Ε, το μεγαλύτερο τμήμα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και περίπου λίγο παραπάνω είναι το προσωπικό, πρώην προσωπικό που αυτή τη στιγμή έχει μία σύνταξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τι θα γίνει λοιπόν με τους ενεργεία υπαλλήλους. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τέσσερα σενάρια. Δεν είναι το μοντέλο, το, το μοντέλο τρεις γάμοι και μία κηδεία, αλλά ε, τρεις, ε, τρία διαζύγια και ενδεχομένως ε, ένας νέος γάμος. Και αυτό θα σας το παρουσιάσω για να σας πω τι γίνεται από πρακτικής απόψεως. Από θεωρητικής απόψεως όμως η εντύπωση μου είναι ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ή εν πάση περιπτώσει η αρμόδια αρχή έχει τρεις επιλογές στη διάθεσή της βάσει του κανονισμού ε, για το ε, προσωπικό, ε, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να διατηρήσει όχι τους υπαλλήλους αυτούς τους Βρετανούς η πιο βία ε, πιθανότητα είναι βεβαίως η παρέτηση τους, ε, άρθρο 28 και 49 ε, του κανονισμού, αν τα συνδυάσουμε και τα δύο, στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε υπάλληλοι μόνο αν διαμένουμε σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήτρα του άρθρου 49 θα μπορούσε να ισχύσει. Δεν θα μπούμε τώρα στη συζήτηση, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα θέμα ερμηνείας, είναι υποχρέωση είναι μία πιθανότητα. Ε, φαντάζομαι ότι είναι μία πιθανότητα, αλλά το ζήτημα παραμένει εκρεμές. Ό,τι και να γίνει υπάρχουν κάποιοι όροι που, πρέπουν, που πρέπει να γίνουν σεβαστοί σε σχέση με την αφαρμογή της διάταξης αυτής. Όχι μόνο δηλαδή πρέπει να ακούσουμε έναν προς έναν τους ενδιαφερομένους, αλλά μετά θα πρέπει να υπάρχει και μία αιτιολογημένη άποψη της αρμόδιας αρχής. Δεύτερη επιλογή πριν περάσω στη δεύτερη επιλογή μάλλον, καλύτερα να διευκρινίσω ότι υπάρχουν πάντοτε διάφοροι διακανονισμοί και πιθανές ε, εξαιρέσεις. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ε, διορίσει ε, έναν μη διαμένοντα σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπάλληλο. Έχουμε βρει δηλαδή στην ομολογία τέτοιου είδους περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι που δεν διαμένουν σε κράτος μέλος της Ένωσης μπορεί να διοριστεί ως υπάλληλο αυτής. Ε, θα μπορούσε λοιπόν πάντοτε να αποτελεί μια πιθανότητα να υπάρξει μια ρήτρα ή ένα συγκεκριμένο ειδικό κεφάλαιο στην Συμφωνία Αποχώρηση σε βάση του άρθρου 50 ε, για να υπάρξει η διατήρηση των Βρετανών υπαλλήλων, εν πάση περιπτώσει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, όλα αυτά είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης κατά την άποψή μου. Να συνεχίσω με τη δεύτερη εναλλακτική επιλογή ε, των πιθανών σεναρίων ε, είναι μια άδεια προ όφελο τη υπηρεσία, κάτι το οποίο προέρχεται από την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού ε, για το προσωπικό, κάτι το οποίο ψηφίσατε το 2013. Ε, όμως η όρη είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι το άρθρο 42 υπάρχει ένας όρος να αποδειχθεί ότι υπάρχουν ανάγκες οργάνωσης ε, συνδεδεμένες με νέες αρμοδιότητες για παράδειγμα που ε, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν ε, νέοι υπάλληλοι και ε, γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ε, αυτή η ειδική άδεια για κάποιους υπαλλήλου. Ε, η νομιμότητα αυτής της διάταξης είναι συζητήσιμη. Έχω βρει τουλάχιστον τρεις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου για το θέμα της νομιμότητας της συγκεκριμένης διάταξης. Και μια τρίτη επιλογή είναι η πάυση από την εργασία ε, χάρη για λόγους υπηρεσίας. Ε, είναι κάτι βέβαια δηλαδή το οποίο επαφίεται στους γενικούς διευθυντές ή στον γενικό διευθυντή. Ε, δεν αποκλείεται όμως σε, κάποια πιο, σε κάποιο πολιτικό πλαίσιο να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιλογή. Όσον αφορά το νέο γάμο που ανέφερα προηγουμένως, το σχέδιο Β δηλαδή, είναι η πιθανότητα που πάντοτε παραμένει ο υπάλληλος ε, ε, ο υπάλληλο των θεσμικών οργάνων ή των υπολείπων ε, υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θελήσει να σεβαστεί αυτά που προβλέπει το άρθρο 50 για τους, για τους ε, συνταξιούχους λογικά δεν θα πρέπει να υπάρχει άμεσος αντίκτυπος ε, γιατί ε, ένας συνταξιούχος έχει υπηρετήσει ήδη ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς έχει δικαίωμα σε σύνταξη αν βεβαίως σέβεστε τους όρους συνταξιοδότησης δεν επεκτείνομαι από αυτού. Όμως το ερώτημα που μπορεί να τεθεί εμέσως πλέον είναι η αηφορία του συστήματος συνταξιοδότησης, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στο σύστημα συλλογικής εξασφάλισης των ε, συντάξεων, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο και εκείνο έχει κάποιες ευθύνες για την ε, εξασφάλιση του συστήματος αυτού. Στο πλαίσιο λοιπόν του προϋπολογισμού θα υπάρξει συνεχιζόμενη χρηματοδότηση του σχετικού προϋπολογισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο το ζήτημα ε, παραμένει εκρεμές. Τώρα, είχε γίνει στην ε, περίπτωση της ε, Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, είχε προβλεφθεί ένα συνταξιοδοτικό ταμείο ad hoc, του οποίου η διαχείριση στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, ε, είχε αποτελέσει μετά ένα δευτερεύον ταμείο της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τότε. Υπήρχαν λοιπόν κάποια προνόμια σε σχέση με την φορολογική μεταχείριση αυτών των συντάξεων. Τελευταία πτυχή που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε είναι ε, η τύχη των υπολείπων που δεν είναι Βρετανοί ε, υπήκουοι, όμως ε, παρόλα αυτά δουλεύουν, εργάζονται για υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή που εργάζονται για υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όλους τους υπόλοιπους υπαλληλου που ε, εργάζονται για μέλη, ε, για Βρετανούς υπαλλήλους ε, άλλων ε, οργάνων. Υπάρχει λοιπόν το θέμα αυτό, αν κατάλαβα καλά διαβάζοντας το έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε εχθές για το οικονομικό καθεστώς του Brexit, το οποίο δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πτυχή που έχει να κάνει με τη μετακόμιση των υπηρεσιών έχει προβλεφθεί. Επίσης εντός του κειμένου αυτού που χθες δημοσιεύθηκε ε, υπάρχει μία πτυχή που αφορά τις συντάξεις, αλλά συμπερασματικά θα ήθελα να σας πω ότι ε, παραμένει το γεγονός ότι όλα θα, θα, θα εξαρτηθούν από τη συμφωνία αποχώρησης. Μπορεί να είναι λίγο απεσιόδοξο αυτό που λέω. Ε, παρόλα αυτά, για να είμαστε αισιόδοξοι, όπως, αν υπάρχει πολιτική βούληση, όπως είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι προηγουμένως, δεν... Ε, Υπάρχει λόγος να μην βρούμε αυτό το ανοιχτό πνεύμα ε, διατήρησης των Βρετανών υπαλλήπων και του ε, λοιπού προσωπικού εντός της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Ήταν και η τελευταία παρουσίαση αυτή. Έχουμε κάποια λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις αν το επιθυμείτε. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, δεν θα απαντήσω άμεσα σε κάποια ερώτηση, αλλά μου κάνατε εσείς νωρίτερα μια ερώτηση και θα ήθελα να απαντήσω τα εξής. Το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου περιέχει διατάξεις που οδηγούν σε προσφυγές στα δικαστήρια. Πρόκειται για θέματα συνταγματικότητας, υποχρεώσεις, θέματα συνταγματικότητας οι γενικές γραμμές. Μια σύντομη λοιπόν απάντηση που θα μπορούσα να δώσω στην ερώτηση που μου κάνατε είναι ότι εξαρτάται ε, βεβαίως κατά πόσο αυτές οι εξουσίες και αρμοδιότητες θα αλλάξουν. Η απάντηση είναι σαφώς ναι. Το Κοινοβούλιο της Σκοτίας σίγουρα θα περάσει από κάποιες μεταρρυθμίσεις. Το θέμα της συνταγματικότητας είναι κάτι που εξελίσσεται Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε από εδώ και πέρα τι θα πρέπει να εκδικάζεται στα δικαστήρια και τα θέματα που άπτονται της συνταγματικότητας από εδώ και πέρα που θα απευθυνόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν μίλησα για αρμοδιότητες, αλλά για το κατά πόσο συνάδουν και συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο. Για τις τεχνίες, αν κατάλαβα καλά, δεν εξηγήθηκε το ότι θα γίνει κύριος από το Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης λέγεται ότι η Ιταλία ενδιαφέρεται και εκείνη να αποφασίσει σχετικά και να έχουμε τέλος πάντων αυτό το τμήμα του δικαστηρίου στο Λονδίνο με την κύρωση της συνθήκης από το Λονδίνο. Αλλά θέλω να ρωτήσω, τι λέει για την γνωμοδότηση 109 ο εισηγητής. Μια που αναφέρεται ότι μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετάσχουν. Τι ερμηνεία μπορεί να δοθεί σε αυτή τη διάδεξη της συνθήκης. για την Ιταλία. Λέει ο συγητής. Αυτό αναείδε στην αρχή της ενισχυμένης εργασίας. Δεν ήθελε η Ιταλία να συμμετάσχει στο ενιαίο σύστημα των ευρωσταχνιών. Άλλαξε όμως την τοποθέτησή της έκτοτε. Όπως είπα και στην εισήγησή μου, θεωρώ ότι υπάρχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Θα ωφεληθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με το που θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Οπότε καλύπτεται και η Ιταλία. Και όσον αφορά την γνωμοδότηση 109, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει κατά δύο τρόπους τη γνωμοδότηση. Πρώτα-πρώτα, αυτό το οποίο ήταν η ερμηνεία η αρχική της Κομισιόν, ότι το ενιαίο δικαστήριο μπορεί να είναι δικαστήριο μόνο για τα κράτη-μέλη. Όμως αν κανείς ε, κολλήσει στο, στο γράμμα της νομοδότησης δεν λέει κάτι τέτοιο. Η νομοδότηση λέει ότι τα κράτη των κρατών μελών ε, θα πρέπει να ενεργούν με σεβασμό στο κοινωτικό δίκαιο. Δεν λέει ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο δικαστήριο μόνο κράτη-μέλη. Οπότε γι' αυτό και το συμπέρασμά μου είναι ότι μια από τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Θα πρέπει το δικαστήριο να γνωμοδοτήσει και να ερμηνεύσει την τοποθέτησή του. Ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κρόαση όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι μια κυρίαρχη απόφαση. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την απόφαση και πρόκειται για την ελευθερία του κάθε λαού να αμφισβητήσει συμφωνίες και προσχωρήσεις. Ευχαριστώ τους ε, οργανωτές γιατί βέβαια εδώ αν κοιτάξω αυτήν την ε, αφίσα βλέπουμε μια χειραψία μεταξύ Βρετανών και Ευρωπαίων. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι πρέπει να δούμε την αποχώρηση του μεγάλου του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι σαν καταστροφή. Οι δύο τελευταίοι ομιλητές μας έδειξαν ότι μπορεί να υπάρξουν λύσεις και ο κύριος Μάθιος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά και ο κύριος Ροντίγκης όσον αφορά τους υπαλλήλους που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Νομίζω δεν αναπτύξατε αρκετά το εναλλακτικό σχέδιο ε, μιλήσατε για την επιλογή εναλλακτική παριθμών 4, δηλαδή μιλήσατε για επανένωση ή ε, νέο γάμο. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε λίγο. Ναι, κοιτάξτε, μιλήσα για νέο γάμο γιατί θεώρησα ότι πρόκειται για την επιλογή μιας άλλης υπηκότητας. Δηλαδή ένας Βρετανός υπάλληλο, ο οποίο θέλει να γίνει Βέλγος, γιατί μένει στο Βέλγιο, είτε τη γαλλική υπηκότητα, γιατί η σύζυγός του είναι Γαλλίδα. Πρόκειται για συγκεκριμένες πραγματικές περιπτώσεις που υφίστανται. Κανείς δεν τους εμποδίζει να επιλέξουν αυτήν την υπηκότητα. Θα πρέπει βεβαίως να δεχθούν όλες τις ε, προϋποθέσεις και τους όρους για την απόκτηση αυτής της υπηκότητας. Κατά την άποψή μου δεν αλλάζει τίποτα ως προς αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους να ζητούν το λόγο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο είδαμε λίγο πιο καθαρά τι μας περιμένει. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας παρουσιάσατε κάποιες από τις δυσκολίες. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ σε αυτή την ακρόαση.